Bien, mes chers collègues, je vous invite à Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Και πριν υποδεχθούμε και τους συναδέλφους Κλοντ Μωράης και Ινκεμποκ, για αυτή την κοινή μας συνεδρίαση, καθώς επίσης και τον Γενικό Διευθυντή ε, της Ακτοφυλακής Συνοριοφυλακής θα ήθελα να σας ε, πω δύο λόγια όσον αφορά πρακτικά ζητήματα τα οποία αφορούν την ε, Επιτροπή μας. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, θεωρώ ότι έχω, έχει εγκριθεί η ημερήσια διάταξη. Να σας πω ότι η έκθεσή μου για το Brexit ε, έχει αναβληθεί, περιμένοντας ε, και την απόφαση του Συμβουλίου ε, και μια έκτακτη συνεδρία θα λάβει η χώρα στις 11 Απριλίου την επόμενη Πέμπτη το πρωί. Αλλά για την ώρα... Δεν είμαι σε θέση να σας πω αν όντω θα λάβει χώρα αυτή η συνεδρίαση, δηλαδή όλα θα εξαρτηθούν από την ε, συνάντηση της διάσκεψης κορυφής δηλαδή που θα λάβει χώρα ε, λίγο πριν και τις αποφάσεις οι οποίες θα έχουν ληφθεί και από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, για την ε, τωρινή μας συνεδρίαση, απλουστευμένη διαδικασία βάσει του άρθρου 50 ε, για το σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και για την αύξηση του κεφαλαίου από την Ρουμανία και την Πολωνία μετά από το Brexit. Το σημείο θα μας απασχολήσει αύριο από τον μόνιμο εισηγητή. Projet préparé par EDER a Τέλος να σας πω ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτρο... μάλλον η τελευταία ε, της Επιτροπής Προπολογισμών θα λάβει χρόνο την Τετάρτη και θα ασχοληθεί με το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2020 καθώς επίσης και τους προϋπολογισμούς που θα έχουν εγκριθεί μέχρι τότε για το 2019 από τον Επιτροπό Ότιγκερ στο τέλος της ε, εν λόγω συνεδρίας της 5ης Ιουνίου. Ε, Καλείστε όλοι ε, σε ένα κοκτέιλ τέλους θητείας έτσι ώστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτά τα πέντε χρόνια συνεργασίας και αμοιβαία κατανόησης προς το συμφέρον πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα σχετικά στοιχεία θα σας ταλούν. Τέλος, λάβατε ανακοίνωση των ε, πρακτικών της συνεδριάσης της 7ης Μαρτίου της 18ης Μαρτίου και της 25ης ε, Μαρτίου. Φαντάζομαι ότι τα διαβάσατε με πολύ μεγάλη προσοχή ε, και αφού δεν έχετε υποβάλει σχόλια μπορώ να θεωρήσω ότι αυτά τα τρία πρακτικά εγκρίνονται. Σας τα είπα όλα αυτά. Και όπως σας είπα και στην αρχή, εδώ έχουμε μια κοινή συνεδρίαση ε, των Επιτροπών ε, ε, ΛΥΜΠΕ και ΚΟΝΤ, ελέγχου προπολογισμού. Μας δίνει ιδέα αυτή η κοινή συνεδρίαση την πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή και να ανταλλάξουμε απόψεις με τον κύριο Ρουτζέρη της Frontex της, ε, του Οργανισμού Ακτοφυλακής Νοριοφυλακής και κύριε Λετζέρη, αν μου το επιτρέπετε και εσείς, θα δώσω πρώτο το λόγο στον Κλοντ Μωράης. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ και οι συνάδελφοι και η Λετζέρη ε, να σας ευχαριστήσουμε και για την έκθεση που αγγίζαμε στη ΛΥΜΠΕ και την παρακολούθηση που δώσετε εσείς για την απαλλαγή του προϋπολογισμού του 2017. Εμείς καλωσορίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής αυτής και την σημερινή ανταλλαγή απόψεων και η Επιτροπή θέλει να μάθει ε, για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Θέλουμε να καταλάβουμε ποιε είναι οι επιχειρησιακές ε, προκλήσει που αντιμετωπίζει η υπηρεσία σα. Το έχουμε συζητήσει βέβαια και στην Επιτροπή μα, αλλά καλό είναι να συζητηθεί και εδώ στην Επιτροπή Δημοσιονομική και την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Μετά από αυτή τη σύντομη δήλωση σας ξαναδίνω το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι η Frontex συχνά είναι στην καρδιά των δημοσίων συζητήσεων και των ε, ανταλλαγών απόψεών μας εδώ ε, είναι πιθανό άλλωστε στην προεκλογική εκστρατεία που ξεκινάει το θέμα της μετανάστευσης να βρεθεί στην καρδιά των συζητήσεων. Αυτή η υπηρεσία ήταν αντικείμενο και νομοθετικών και δημοσιονομικών διαδικασιών. Εξακολουθεί να μας απασχολεί και στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης της εντολής τη στο επομενο πολιτευθυνο νομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 μας απασχολεί διότι ε, οι πιστώσει στο, στη γραμμή, στο κεφάλαιο 3 ε, του προπολογισμού ε, είναι αυτή τη στιγμή υποσυζήτηση. Προετοιμάζουμε και τον νέο προπολογισμό του 2020. Μας απασχολεί και για την εφαρμογή και τη διαχείριση του προπολογισμού και την απαλλαγή του καθώς και τα ζητήματα ανθρωπίνων πόρων. Ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτημα για αυτές τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, ε, διότι ε, προβλέπεται να ε, προσληφθούν γύρω στους 10.000 υπαλλήλου. Ε, και βεβαίως σε επικοινωνιακό επίπεδο ορισμένε φορές οι συνοριοφύλακες, οι ακτοφύλακες έχουν να αντιμετωπίσουν δραματικές καταστάσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Κύριε Εκτελεστική Διευθυντή, Διευθυντή της Frontex, θέλουμε να σας ακούσουμε για την υπάρχουσα κατάσταση στην υπηρεσία σας, ποια είναι τα σχέδιά σας, ποιες είναι οι δυνατότητες που θα έχετε έτσι ώστε να αυξηθούν ε, οι ανθρώπινοι πόροι σας ε, ε, μέσα σε ποιο προθεσμία πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο να έχει συμβεί αυτό. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεση σας για την παρουσίασή σας. Μόλις μοιράστηκε η έκθεση του 2018 στους συναδέλφους εδώ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Merci, le Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις επιτροπές προεπολογισμού δημοσιονομικού ελέγχου και ΛΥΜΠΕ που μου δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσω εδώ τη δραστηριότητα της υπηρεσίας μας. Θα ξεκινήσω με κάποια επιχειρησιακά στοιχεία και θα μιλήσω και για την μετατροπή της, τους κινδύνους αλλά και τις προκλήσεις που συνοδεύουν αυτήν την αλλαγή και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την διοικητική διακυβέρνηση, ε, την εσωτερική που αφορά βεβαίω σίγουρα την Επιτροπή Προπολογισμού και την Επιτροπή του Ελέγχου. Και θα ήθελα να αναφερθώ επίση και στην ευθύνη απέναντι στο Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τα, επιχειρησιακά επιτεύγματά μα, η έκθεση του 2018 που μοιράστηκε σα επιτρέπει να δείτε το μέγεθο των ε, δραστηριοτήτων μα. 11.000 ε, ε, συνοριοφύλακες συμμετείχαν σε αναπτύξεις της υπηρεσίας Frontex εντός του 2018 θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 τα δύο-τρία τελευταία χρόνια η Frontex πραγματικά ε, έχει γίνει μια υπηρεσία συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων ε, υπάρχουν 21 πλοία που αναπτύσσονται καθημερινά 345, 445 πτήσεις επιστροφής για άτομα που διαμένουν παράτυπα στην Ένωση, τέσσερις φορές δηλαδή περισσότερες απομακρύνσεις από το 2016. Το 2018 είχαμε 12.500 απομακρύνσεις παράτυπων μεταναστών, 4.000 νορφύλακες και ακτοφύλακες ε, καταρτίστηκαν ε, ε, το 2018 τριπλά, το τριπλάσιο αριθμό από ό,τι στο παρελθόν, 11 αξιωματικοί σύνδεσμοι στα κράτη-μέλη. ο δεύτερο κύκλος ε, της ε, έρευνας ευαλωτότητας ολοκληρώνεται και πλέον από από στις τρίτες χώρες ετοιμάζουμε μια επιχείρηση που θα ξεκινήσει στα Δυτικά Βαλκάνια την άνοιξη του 2019. Επίσης ε, έχουμε επεκτείνει τις επιχειρήσεις μας και στην Αφρική στα πλαίσια παραδείγματο χάρη των αξιωματικών συνδέσμων στον Νίγηρα. Έχουμε πολύ καλέ συζητήσει και με την Αίγυπτο και με τη Σενεγάλη. Ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και ένα νέο οικονομικό σχήμα ε, έχει προβλεφθεί έτσι ώστε να απλουστευτεί ε, η διακυβέρνηση στα πλαίσια της ε, υπηρεσίας. Ε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια διοικητικής ε, απλούστευσης ε, με αποτέλεσμα από τις χίλιες πράξεις να έχουμε φτάσει στις 400. Έγινε λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και βεβαίως προσπαθούμε έτσι ώστε όλες αυτές οι αλλαγές να ακολουθούν σωστά από το προσωπικό. Μπορώ να πω σε αυτό το στάδιο ότι δεν είμαστε πλέον σαν τους πυροσβέστες που προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές το καλοκαίρι, αλλά είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε ε, σύγχρονες δομές ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2015 έχει αυξήσει κατά 3,5 φορές ε, το ε, μέγεθος των, της προσπάθειάς τους. Και τώρα να σας εξηγήσω λίγο παραπάνω τι γίνεται με την μεταρρύθμιση τη υπηρεσία που ξεκίνησε το 2015-2016. Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε στη νέα εντολή της. Ε, επέδειξε λοιπόν η ηγεσία και οικοδόμησε μια ισχυρή βάση στην οργάνωση και ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στην ταχεία ανάπτυξη. Και έτσι είχαμε νέους ε, διευθυντές και έτσι δημιουργήθηκε μια πολύ δεσμευμένη διευθυντική ομάδα και ένα ηγετικό πρόγραμμα καταρτίστηκε για την διεύθυνση, νέες αξίες, μεταξύ των οποίων και η λογοδοσία. Η υπηρεσία λοιπόν πέρασε μια βαθιά μεταρρύθμιση με τον σχετικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσαρμόσαμε λοιπόν τον εσωτερικό κανονισμό και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ε, νέας διευθυντικής ομάδας και έτσι η υπηρεσία μας κατάφερε να ανταπεξέλθει σε όλες τις πτυχές της νέας εντολής. Αντιλαμβάνομαι τη μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε ακόμα μπροστά μας και σκοπός μου είναι να συνεχίσω στο ίδιο πνεύμα για τις μελλοντικέ ε, μεταρρυθμίσεις. Η αύξηση του προπολογισμού συνοδεύτηκε από διαρκή αναζήτηση για αποτελεσματικότητα και αποβατικότητα και έτσι η παρακολούθηση, για παράδειγμα, της ε, χρήσης των πόρων αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του πώς μπορούμε να παρακολουθούμε την επίτευξη των στόχων. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό έγκλημα στην ε, γειτονία της Ευρώπης. Και η μεταρρύθμιση της σχετικής ε, διευθυντικής εικόνας ήταν βασικό μέλημά μας. Εξετάσαμε την απόδοση εξετάσαμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης μιας ε, αποτελεσματικής ε, διαχείρισης ε, και με ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και λογοδοσίας, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Το νέο σύστημα αντιπροσωπιών και υποαντιπροσωπιών, για παράδειγμα, αποφασίστηκε και εγώ εφάρμοσα ένα σύστημα το οποίο προσωμιάζει με αυτά που προβλέπονται από το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επόμενα χρόνια η υπηρεσία θα λειτουργήσει με προενεργό τρόπο χάρη και στις ενισχυμένες ικανότητές της, όπου ανακύψουν εκτέκτες περιστάσεις. Και όλο και πιο πολύ θα δράσει και ως ε, ομάδα δημιουργίας ε, δυναμικού στα κράτη-μέλη. Φυσικά, μαζί με τι ευκαιρίε έρχονται και κίνδυνοι, γιατί η υπηρεσία λειτουργεί σε ένα πολύ ευαίσθητο περιβάλλον. Η διαχείριση των συνόρων δεν αποτελεί αυτό σκόπο. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή πολιτική και να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα των πολιτών σε τομεί όπω η ασφάλεια, η μετανάστευση και η οικονομική ανάπτυξη. Και για αυτό το λόγο λοιπόν η ενοποιημένη διαχείριση συνόρων αποτελεί τόσο περίπλοκο ζήτημα και η εφαρμογή αυτή είναι μεγάλη πρόκληση και για την υπηρεσία μα, αλλά και για τι αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι Ευρωπαίοι θύνοντες έχουν κατανοήσει καλά το λόγο και το ρόλο τη υπηρεσία μα και την ανάγκη να εφαρμοστεί μια συνεργοφυλακή και ακτοφυλακή όχι μόνο με νομικέ αλλαγέ στην εντολή αλλά με πραγματικέ και ουσιαστικέ αλλαγέ. Και όλε αυτέ οι εξελίξει θα επιτρέψουν και στην υπηρεσία αλλά και στι εθνικέ αρχέ να αντιμετωπίσουν το μέλλον πολύ πιο καλά προετοιμασμένε. Θα υπάρξει μια σταδιακή μετάβαση από την ε, αντίδραση στην ε, προ... των, ε, των προτέρων πρόληψη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των σύνορων. Και ο νέο τρόπο λειτουργία μα θα βασιστεί σε μια ενισχυμένη ευαισθητοποίηση για τι εκάστοτε καταστάσει σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, περιοχές πρώτων συνόρων, όπως Eurosur για παράδειγμα, και βέλτιστη χρήση των στατιστικών στοιχείων από τα στατιστικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα κρίσιμα στοιχεία θα μας βοηθήσουν για τη διαμόρφωση της πολιτικής μας και στη βέλτιστη χρήση των ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενοποιημένη διαχείριση των συνόρων. Αυτό αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα χάσματα και τη ε, υπηρεσία μα αλλά και των αρμόδιων αρχών. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και στα πορίσματα του της αξιολόγησής μας. Θα πρέπει αυτά τα χάσματα λοιπόν να τα κλείσουμε μαζί με την κινητικότητα, για παράδειγμα, μεταξύ των διαφορών α, θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή κουλτούρα, αν θέλετε, και η ταυτότητα εργασίας και η ομοιογένεια ξεπερνάει τα θέματα της ε, στολής, για παράδειγμα. Θα πρέπει να δουλεύουμε με τους ε, ομολόγους μας σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, αντιδρομίας, να υπάρχει μια συντονισμένη ε, προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα κράτη-μέλη για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, για να υποστηριχθούν αυτέ οι διαδικασίε. Θέλουμε να έχουμε ό,τι καλύτερο γίνεται στην ακτοφυλακή και στη συνειδητοφυλακή. του καλύτερου. και μία από τι βασικέ προκλήσει τουλάχιστον για την υπηρεσία, θα είναι να μπορέσει να προσελκύσει ακριβώ αυτό το κατάλληλο προσωπικό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και διάφορε πτυχέ. οικογενειακή κατάσταση, κατεύθυνση, και γενικοί όροι της εργασίας. Θα πρέπει να αναπτύξουμε μια δυναμική ε, εικόνα για να προσελκύσουμε τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους. Να πω δεξής τώρα. Ο σχετικός κανονισμός όχι μόνο επιβεβαιώνει τη λειτουργική εντολή της υπηρεσίας, αλλά δίνει και μια στρατηγική πτυχή στις εργασίες μας. Η υπηρεσία Ανέπτυξε λοιπόν ένα λειτουργικό σύστημα και στρατηγική για την διαχείριση των συνόρων βάσει των ε, νομοθεσιών, ε, νομοθεσιών και της EU IBM. Και όλα αυτά λοιπόν πρέπει, θα πρέπει πλέον να εφαρμοστούν και στις εθνικές ε, στρατηγικές για τη διαχείριση των συνόρων. Η υπηρεσία λοιπόν θα παρακολουθήσει τη διαδικασία αυτή ω θεματοφύλακα τη στρατηγική για την ολοκληρωμένη διαχείριση σύνορων. Αυτή η στρατηγική λοιπόν έχει ένα νέο στόχο να μειώσει την ευαλωτότητά μα και να αυξήσει την ασφάλειά μα και την εύρετη λειτουργία των εξωτερικών σύνορων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξει τι ε, δυνατότητε διατήρηση των σύνορων. Είναι στο πνεύμα τη κοινή ευθύνη. ρόλο λοιπόν τη υπηρεσία θα είναι να συντονίσει, να εφαρμόσει, να αξιολογήσει τι σχετικέ δραστηριότητε και τα σχετικά μέτρα και σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή λοιπόν ε, αξιολόγηση τη ευαλωτότητα προποθέτει να υπάρχει μία πραγματικά έντιμη σχέση σε ό,τι αφορά τώρα το οικονομικό πλαίσιο, το νέο πίδι που έχει αυξήσει τους ε, πόρους ε, για την ενοποιημένη διαχείριση των συνόρων και η υπηρεσία μας θα είναι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή του προτινόμενου προπολογισμού για το νέο ποδοπού θα γίνει αναζητώντας συνέργειες και πλήρη συμπληρωματικότητα με τα εθνικά προγράμματα. Αυτό θα ισχύσει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του υφιστάμενου σώματος με πάνω από 2 δις για την ε, κατεύθυνση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν προωθούμε το σχέδιο ενοποιημένη διαχείριση συνορών που θα λάμβει υπόψη του δύο πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και τη Συνοριοφυλακή, στην υπηρεσία και τι εθνικέ αρχέ. Θα μεγιστοποιήσουμε επίση τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για να υπάρξει πιο ανθεκτική διαχείριση συνόρων και μια μεγάλη επιχείρηση καινοτομία όπου τα καινούργια συστήματα, όπως το αίτια στο σύστημα εξόδου-εισόδου, θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δεν οικοδομούμε το φρούριο της Ευρώπης. Φτιάχνουμε ένα καλά λειτουργόν σύστημα διαχείριση των όρων. Να κλείσω τώρα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο και την λογοδοσία, την διαφάνεια έναντι των Ευρωπαίων πολιτών. Πέρσι συμμετείχα σε τέσσερις ακροάσεις της ΛΥΜΠΕ και επτά άλλες ακροάσεις που διοργανώθηκαν στο Κοινοβούλιο από επιτροπές. Και ξέρω ότι αυτό δεν ε, πρόκειται να μειωθεί στο μέλλον, θα αυξηθεί μάλλον, γιατί ο τρέχον κανονισμό περιλαμβάνει διάφορε διατάξει σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει λογοδοσία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαστε ιδιαίτερα δεσμευμένοι να τηρήσουμε τι προθεσμίε και να ανταποκριθούμε στι υποχρεώσει μα. Πέραν από αυτό, υπάρχει και ο θεσμικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το πολίτε ε, πρόγραμμα εργασία μα και το ετήσιο πρόγραμμα ε, εργασία μα και τη απαλλαγή ε, και τη ετήσια έκθεση. Ανέφερα λοιπόν ακριβώ τη διαφάνεια τη υπηρεσία, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να έχει το κοινό πιο πολλέ πληροφορίε για τη δουλειά μα. Ενημερωμένη λοιπόν περιγραφή των καθηκόντων της υπηρεσίας πλέον διατίθεται στην ιστοσελίδα μας όλες τις επίσημες γλώσσες και επίσης το έργο της υπηρεσίας μας συχνά παρουσιάζεται υπό το πρίσμα των λαφρομεταναστών. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι εργαζόμαστε για τους Ευρωπαίους πολίτες για να εξασφαλίσουμε ότι θα διασφαλίσουμε την, το χώρο ελευθερής μετακίνησης. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πραγματικά δεν είναι κάτι πολύ απτό και η υπηρεσία είναι το λειτουργικό σκέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν από το εξή. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας κάνει ξεκάθαρο ότι χρειάζεται όλο και πιο πολύ λογοδοσία. Υπάρχουν πολλά επίπεδα λογοδοσίας. Καταρχάς, έχουμε το επίπεδο το διευθυντικό του Διοικητικού Συμβουλίου της υπηρεσίας. Έχουμε μια σειρά οικονομικών αρχών, ελεκτικό συνέδριο, διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος Επόπτη ε, Προσωπικών Δεδομένων και σε πολιτικό επίπεδο προφανώς και τα θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο εδώ έχει πολλές αρμοδιότητες ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της υπηρεσία μας και τέλος εσωτερικά η υπηρεσία έχει και εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις το δικαίωμα των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων είναι αυτόνομες ε, θέσεις και έχουμε και ένα εξωτερικό σώμα συμβούλων που δίνει, ε, παρέχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά θέματα που των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αξιότιμοι βουλευτές, η αύξηση των ευρωπαϊκών πόρων για τη συνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή ε, έχει σημαίνει πολλές προσδοκίες και πολλές ε, ευθύνες. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι σαφής σε ό,τι αφορά τη δημοκρατική εξισορρόπηση και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Συνόρων να καλωσορίσω την κυρία Γκρέσλε που μόλις έφτασε. Κύριε Διευθυντά, με την παρουσίασή σας ήδη απαντήσετε κάποια ερωτήματα, αλλά θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Ολμάιερ της, της ομάδας προπολογισμού, της επιτρέψης Προϋπολογισμού και εισηγήτριας για τον ε, προϋπολογισμό του 2020. Είναι ο κύριος Γκέγερ που είναι ο μόνιμος εισηγητής μας για τις υπηρεσίες και στη συνέχεια θα απευθυνθώ σε εσά κυρία Γκρέσλε και προς τον κύριο Μωράες έτσι ώστε και εσείς να μας πείτε ποιος από εσά θα θέσει ερωτήματα ε, ή παρατηρήσεις ε, προς τον ε, κύριο Λετζέρη. Κυρία Ολμάιερ. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεζουρή, καλώ ορίσατε στην Επιτροπή μα και χαίρομαι που μα παρουσιάσατε την έκθεσή σα με πολύ ακριβή αριθμητικά στοιχεία και μάλιστα με πολύ συνοπτικό τρόπο. Αυτό που θα με ενδιαφέρει είναι το εξή ε, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό του 2020 και για του επόμενου προπολογισμού. Θα υπάρξει αύξηση των πόρων της Frontex και η Frontex στην παρούσα φάση προσανατολίζεται όχι τόσο πολύ όσο ένας μηχανισμός αντιμετώπισης εκτακτών κρίσεων πλέον, ως, όσο ως μια διαρκή παρουσία πλέον στα κράτη-μέλη. Ανακύπτει λοιπόν το εξή ερώτημα. Κατά το παρελθόν είχαμε προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, έγκυρη κινητοποίηση των δυνάμεων. Κατά δεύτερον, Δυνάμει οι οποίε έπρεπε να προσληφθούν επί τόπου, έπρεπε να προσληφθούν αρκετά γρήγορα. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσει να σα θέσω. Καταρχάς, αρκούν τα ειδικητικά σας στελέχη προκειμένου να το επεξέλθουν στις ανάγκες σας. Κατά δεύτερον, οι μισθοί αρκούν για να μπορέσουμε να έχουμε ε, έμπειρους, έμπειρο ε, προσωπικό στη Frontex και όχι μόνο νεαρούς ε, εκπαιδευόμενους, γιατί ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε από πλευρά προπολογισμού αυτό. Κατά τρίτον, σε ό,τι αφορά το θέμα της αποτελεσματικότητας, τα κράτη-μέλη στα οποία δραστηριοποιείστε είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά τη συνεργασία ή εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα. Σε κάποιε περιπτώσει, δηλαδή προσπαθεί κάποιο κράτος να κρατήσει λίγο μακριά τη Frontex, ε, απ' έξω. Γιατί ενδεχομένω κάποια κρατημέλη να έχουν συμφέρον να μην ε, γνωρίζει η Frontex κάποια πράγματα και δεν επιτρέπεται ε, πρόσβαση στη Frontex σε κάποια μέρη. Και αυτό θεωρώ ότι ρυθμίζεται με τον νέο κανονισμό. Κατά τα άλλα, να σας ευχαριστήσω και για την καλή φήμη που έχει η Frontex στο κοινό, στους πολίτες της Ευρώπης. Το λέω αυτό ξεκάθαρα γιατί πιστεύω ότι συνολικά και η εκπαίδευση και ο τρόπος επέμβασής σας δημιουργεί πραγματικά θετικές εντυπώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ Μόνικα. Θέλετε να απαντήσετε ε, αμέσως και αν είναι δυνατόν ε, σύντομα στις ερωτήσεις της κυρίας είναι σαφές ότι οι ικανότητες διαχείρισης της υπηρεσίας πρέπει να ενισχυθούν και αυτό πραγματικά αποτελεί ένα το μεγάλο στόχος μου, από τους μεγάλους στόχους Για παράδειγμα, η στρατηγική ICT. Αυτό χρειάζεται. Επίσης, όπως διευκρίνησα, θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί στις διαδικασίες μας. Επίσης, προσλάβαμε καινούργιο προσωπικό Και προφανώς ε, προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε τα, τους επόμενους μήνες. Κατά πόσον τώρα μπορούμε να προσλάβουμε έμπειρους συναδέλφου. Ε, συναδέλφους. Εδώ έχουμε λίγο κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά το συντελεστή διόρθωση και θα πρέπει να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά προφανώς και στόχος μου είναι να συνεργαστώ στενά με τις ε, εθνικές αρχές προκειμένου στην τελική ανάλυση να μην δρούμε ανταγωνιστικά μεταξύ μας, αλλά να μας βοηθήσουν. Να υπάρξει μια συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, προστασίας των σύνορων. Κατά πόσο μας ε, στερούν την πρόσβαση σε προβληματικές περιοχές τώρα, κάποια κρατημέλη. Έχουμε καλύτερη γενικά εικόνα σε ό,τι αφορά την ανάλυση δηλαδή των ευαίσθητων σημείων που έχει ήδη γίνει, είχε μεγάλα αποτελέσματα, αλλά προφανώ μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρο, κ. Γκάιερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώ ορίσατε και από πλευρά μα. Βλέπετε λοιπόν τι απασχολεί την Επιτροπή μα, γιατί προ την ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν και οι δικέ μου ερωτήσει. Η πολιτική γενικά έχει την τάση να θέλει να εφαρμοστούν γρήγορα γρήγορα οι αποφάσεις. Αποφασίστηκε λοιπόν ένας ανώτατος αριθμός 10.000 υπαλλήλων και οι πολιτικοί θεωρούν ότι αυτό μπορεί αύριο μεθαύριο να έχει εφαρμοστεί. Αυτό που με απασχολεί εμένα είναι σε σχέση με αυτά που έθεσε και ως ερώτημα η κυρία Χολμάιερ. Εσείς πού βρίσκεστε σε ό,τι αφορά το διοικητικό σκέλος, σε τι χρονοδιάγραμμα θέλετε ότι μπορείτε να δράσετε θα υπάρξει κάποια αναβολή στην υλοποίηση των ηλεμένων αποφάσεων λόγω των προβλημάτων που αναφέρατε με τον συντελεστή προσαρμογής σε, ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους υπαλλήλου. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Και τα δεύτερον, στην επιστολή προς τον Πρόεδρο Μωράες μιλάσατε, μιλήσατε για βασικούς δείκτες μεταρρυθμίσεων. Key Performance Indicators. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς εννοείται με αυτόν τον όρο. Ωραία, αν είναι δυνατόν επίσης πολύ σύντομα να απαντήσετε ε, μία ακόμα φορά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες προκαταρτικές διαβουλεύσεις και για να προσληφθεί αυτό ο μεγάλο αριθμό προσωπικού, θα πρέπει να συνεργαστούμε για τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμό. Και εδώ πρέπει να σα πω ότι έχουμε διάφορε ιστορικέ διαβουλεύσει για την ε, δομή τη ε, υπηρεσία. Είναι σαφή η δομή τη υπηρεσία. Έχουμε τι 14 ε, υπηρεσίε. Έχουμε προετοιμαστεί λοιπόν σε επίπεδο Frontex. Τώρα φυσικά πρέπει να συζητήσουμε και το χρονοδιάγραμμα των συγκεκριμένων με τα κρατημέλη. Και πιστεύω ότι στο σημείο αυτό πρέπει σκοπός μας να είναι να προσλάβουμε έμπειρους συνοριοφυλακές. Εδώ αυτό θα πρέπει να αποτελέσει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στόχο μας. Αλλά φυσικά να προσλάβουμε και νεαρούς, προκειμένου να τους εκπαιδεύσουμε εμείς και να μάθουν σε εμά τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή ενδεχομένω να εργαστούν κάποια χρόνια και στις εθνικές υπηρεσίε και μετά να επανέλθουν στην ε, Frontex. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε όμως με τα κράτη-μέλη. Μπορούμε ασφάλως να ξεκινήσουμε πάρα αυτά. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να είχαμε και λίγο παραπάνω χρόνο να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι μέχρι το 2027 έχουμε ένα στόχο τον οποίο θα πρέπει να έχουμε πετύχει και προφανώς αυτό δεν το ξεχνάμε σε ό,τι αφορά αυτούς τους βασικούς δείκτες απόδοσης Key Performance Indicators. Να πω το εξής. μα κάνουμε μια αξιολόγηση του είδους επιχειρήσεων και ενδεχομένως να χρειαστεί να τροποποιήσουμε κάπως το είδος παρεμβάσεών μας. Έχουμε λοιπόν κάποιους δείκτες κλειδί για την απόδοση που προσμετρούν το κατά πόσον οι εθνικές αρχές χρησιμοποιούν και εκτιμούν τις υπηρεσίες μας. Αυτό για παράδειγμα αποτελεί ένα βασικό δείκτη απόδοσης. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα το λέγω να δώσω στην Πρόεδρο την κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λετζερή και ζητώ συγγνώμη που σας ε, Έχασα λίγο την αρχή και σας παρουσίαση. Σας σκεφτόμουν πολύ το Σαββατοκυριακό. Στα γερμανικά συνδικάτα συζητούσαμε το θέμα της Frontex και... Ανέκυψε το θέμα της προστασίας και της διάσωσης των μεταναστών. Έχετε σώσει πιο πολλούς από ό,τι έχετε επιστρέψει. Και εδώ λοιπόν τι το θέμα. Το θέμα του συντελεστή Βαρσοβίας. Ε, συντελεστής Λουξεμβούργου θα ήταν καλύτερος προφανώς, αλλά αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει ένα πρόβλημα, γιατί οι υπάλληλοι δεν εργάζονται στην Βαρσοβία. Είναι αριθμητικό στοιχείο αυτό για άτομα τα οποία εργάζονται κάπου αλλού. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσε να επιληθεί με πολύ ευλογό τρόπο για σε κανονικές συνθήκες. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει τέτοιο θέμα. Και ύστερα, οι 10.000 αυτές οι θέσεις, τις οποίες ακούμε ξανά και ξανά. Πείτε μας, τι κοστίζει κάθε θέση. Και μάλιστα το συνολικό κόστος, όχι τα επιμέρους κόστη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, σώζουμε μετανάστες, σώζουμε ανθρώπους ασφαλώς. Ε, ξέρετε τα αριθμητικά στοιχεία. Στα πλαίσια όμως της συνοριαφυλακής και κυρίως στη Μεσόγειο, στην Κεντρική Μεσόγειο και στην Ελλάδα και στην Ισπανία, διασώσαμε 36.000 μετανάστες το περσινό έτος. Το 2016 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 90.000 μετανάστες. Είναι καθήκον μας. Και δουλειά μας. Αυτό σημαίνει όταν χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις μας στα πλαίσια της νοριαφυλακής. Σε ό,τι αφορά τώρα τον συντελεστή προσαρμογής και διορθώσεις θα έχουμε διάφορες εθνικότητες υπαλλήλων. Έχουμε τους υπαλλήλους που θα είναι στην Βαρσοβία, αλλά αυτή θα είναι μια μειοψηφία, μειονότητα. 700 υπάλληλοι. 10% των υπαλλήλων μας. Αυτό που θα πρέπει να ρυθμίσουμε και προφανώ θα πρέπει να βρούμε στην κατεύθυνση αυτή τα κατάλληλα συστήματα υπολογισμού. Αυτό που πρέπει να ρυθμίσουμε λοιπόν είναι να διατηρήσουμε ευελιξία. Να διατηρήσουμε τη δυνατότητα, αν για παράδειγμα χρησιμοποιούμε στην και στη Βουλγαρία ή στο αεροδρόμιο της ε, Στοκόλμης. Πώς μπορούμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό, αν αυτή είναι η ανάγκη που έχουμε. Σήμερα δεν έχω κάποια απάντηση να δώσω στο ερώτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να σκεφτούμε και κάτι παραπάνω από το συντελεστή ε, προσαρμογή ε, της έδρας. Σε ό,τι αφορά το κόστος, το πόσο κοστίζουν 10.000 συνοριοφυλακές. Δεν το έχουμε υπολογίσει. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Αλλά θα το δούμε συνολικά και θα το συμπεριλάβουμε σε μια έκθεση σε ό,τι αφορά για παράδειγμα και τον εξοπλισμό, γιατί αυτοί οι υπάλληλοι θα έχουν το δικό τους εξοπλισμό. τι συσκευέ, για παράδειγμα, που χρειάζονται στην εργασία του, τα αυτοκίνητά του, θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αεροπλάνα χωρίς να επιβαρύνουμε τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για ένα συνολικό λοιπόν πακέτο και το οποίο θα πρέπει να υπολογιστεί. Ελπίζω του χρόνου να είμαι σε θέση να σα δώσω μία απάντηση. Αυτό που με ενοχλεί χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Στον τομέα των εξωτερικών της υπηρεσιών, μάλλον στις ε, σε ό,τι αφορά σχέσει, ε, αυτό θα αντιστοιχούσε, 10.000 θέσει αντιστοιχούσαν σε 2 δι. Αλλά πιστεύω ότι δεν επιτρέπεται να μην ξέρουμε γιατί αριθμητικά στοιχεία μιλάμε. Si Εάν ήταν ε, το μισά, θα κόστιζε ένα δις το χρόνο. Κλοντ um, um, uh, Άκουσα την κυρία Γκρέσσες που ε, σχολίασε τον ρόλο της ε, Frontex. Εγώ να πω ότι έλειπε ένα στοιχείο όντω εδώ, ε, ε, γιατί πρέπει να σας πω ότι Αύριο θα εγκρίνουμε την αναθεώρηση του Frontex. Ε, πρόκειται για μια ε, πρόταση που αφορά 10.000 ε, υπαλλήλους και πραγματικά τραβάει το βλέμμα των εξωτερικών ας πούμε ανθρώπων αλλά παρόλα αυτά είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη σκοπιά αυτών που είπε η κυρία Γκρέσσερ προηγουμένως. Είναι όντως πολύ σημαντική η δουλειά της Frontex. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όμως και πόσες είναι οι προσδοκίες που έχουμε τα εξωτερικά σύνορα είναι όντως ε, πολύ ε, ευραία, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποιους ε, δείκτες σε σχέση και με την δυσκολία του έργου της υπηρεσίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε σε κοινέ συναντήσεις με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και Ελέγχου του Προϋπολογισμού ακριβώς περί τίνος πρόκειται, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα έχουν τα πράγματα. Μία συνάντηση σαν τη σημερινή είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά. Ε, και ο κύριος Γκάγερ και η κυρία Χολμάγερ, η κυρία Γκρέσλερ ε, έχουν πολύ, παρακολουθούν με πολύ μεγάλη προσοχή όλα αυτά τα θέματα εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Το είπαν άλλωστε και όλοι οι προλαλήσαντες. Εσείς βέβαια απαντήσατε πάντα με πολύ θετικό πρόσημο αλλά υπάρχουν και όλα τα στοιχεία τα οποία εμείς είχαμε αναφέρει σε μια επιστολή ε, τα ανέφερε και η κυρία Χολμάγερ. Ο κύριος ε, Γκάγερ επίσης ε, μας είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και τα άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μαζί μου, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα έχουν τα πράγματα και στο επόμενο πεί. Δεν μπορεί να υπάρξουν περικοπές, γιατί εσείς θα έχετε σαν υπηρεσία πολύ μεγαλύτερες ανάγκες. Θέλω λοιπόν ε, να υπογραμμίσω τρία σημεία τα οποία ήδη συνάδελφοι ε, έχουν αναφέρει. Πώς καλύπτονται οι υψηλές θέσεις, ε, η διαφάνεια, δεν το λέω επικριτικά, απλώς είναι ένα θέμα καλύτερης κατανόησης, έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Υπάρχουν και κάποια ελάσσονα σημασία σημεία, τα οποία δεν είναι τόσο σημαντικά βέβαια, Έχετε απαντήσει ήδη σε αρκετά θέματα, αλλά δεν ξέρω και αν συμφωνούν οι συνάδελφοι, αλλά ίσως θέλουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Γιατί αύριο θα μας ε, ε, ρωτάνε, ναι, 10.000, είναι πολλές οι 10.000, ε, άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που θα μας θέσουν. Σύντομα, αν μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν ξεκινήσαμε αυτήν την αξιολόγηση ευαλωτότητα ε, στα κράτη-μέλη τη Ένωση, τα μισά κράτη-μέλη δεν ήξεραν ποιο ήταν το κόστο τη διαχείριση των συνόρων. Για να είμαι ειλικρινή, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν κάτι θέλουν να κρύψουν. Απλά δεν θέλουν να απαντήσουν. Όμως, ε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα ε, ε, όταν μου εξήγησαν ε, το γιατί δεν, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν το σώμα των 10.000 συνοριοφυλάκων θα παίξει ένα ρόλο μόχλευσης ε, για τον εξυγχρονισμό και τη δημιουργία ουσιαστικά μιας σύγχρονης δυνατότητας φλέξης των συνόρων που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και που χρειάζονται τα κράτη-μέλη. Όχι για να, να επαναλάβουμε απλά αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, αλλά και για να προετοιμάσουμε ενεργά το μέλλον να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή καλύτερα τις νέες τεχνολογίες, να προσπαθήσουμε ε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να είμαστε πιο ευέλικτοι. Το, το θέμα κλειδί εδώ, το κλειδί εδώ είναι η ευελιξία, να μπορούμε να αναπτύξουμε γρήγορα αυτούς τους 10.000 ανθρώπους από το ένα μέρος στο άλλο όταν ε, έχουμε κάποια έτσι αύξηση των, των πίεσης ε, ε, υποστηρίζουμε τις Ισπανικές Αρχές τον Ιούνιο, στον Αύγουστο, πούμε, ε, για τους ελέγχους, τους κανονικούς ελέγχους ε, στα πλοία που πάνε από την Ισπανία στο Μαρόκο και επιστρέφουν από εκεί. Ε, διότι γνωρίζουμε ότι εκείνη την εποχή υπάρχει με περισσότερη δουλειά. Και υπάρχουν και άλλε τέτοια, τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με την παράτυπη μετανάστευση και βεβαίω ο ρόλος εδώ είναι να, της ε, υπηρεσίας είναι να εκλοσκοπήσουμε τους ενδιαφερόμενους, ε, να καταγράψουμε τα στοιχεία τους για να προετοιμάσουμε και την επιστροφή αυτών που πρέπει να επιστραφούν. Υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Έχουμε και τη δυνατότητα να διενεργήσουμε ελέγχους ε, μέσω του συστήματος πληροφοριών Schengen. Υπάρχει και το σύστημα αιτίας η υπηρεσία λοιπόν όλο και πιο συχνά θα συμμετάσχει στην καθημερινή εργασία των, της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής και αυτό δεν είναι μόνο η υπηρεσία μας, είναι ένα δίκτυο ουσιαστικά εθνικών αρχών των κρατών μελών και της υπηρεσίας μας. Βεβαίως ό,τι αφορά το κόστος εγώ είμαι πεπισμένος ότι τα επόμενα πέντε χρόνια χρησιμοποιώντα και το νέο πολιτεύσιο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να εξυγχρονίσει τι δυνατότητε που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά σύνορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μα μένει ένα τέταρτο για την ανταλλαγή απόψεων. Έχουν στήσει πολύ τον λόγο. Καλό θα είναι να είστε σύντομοι. Θα ακούσουμε όλε τι ερωτήσει και θα απαντήσει στο τέλο ε, ο συνάδελφο. Η κυρία Σατζεντίνη από την Επιτροπή Λίμπε έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όντως ε, είδαμε με χαρά ε, τον διευθυντή στην ΛΥΜΠ. Έχει έρθει, ε, έχει φορές στην Επιτροπή μας. Κάποιες φορές σας καλέσαμε και δεν μπορείτε να έρθετε βέβαια. Μας στείλατε και μήνυμα ε, μέσω βίντεο μια φορά. Καλύτερα να στέλνετε αντικαταστάτη όμως. Διότι στην επόμενη θητεία το θέμα αυτό σίγουρα θα είναι στην επικαιρότητα και αν δεν μπορείτε να έρθετε εσείς ε, δεν νομίζω ότι αρκεί ένα μήνυμα βιντεοσκοπημένο, έτσι. Ε, εκτιμούμε πάντως που, που ήρθατε, θέλουμε να σας βλέπουμε και πιο συχνά, μπορείτε να στέλνετε κάποιον άλλον, αν δεν μπορείτε εσείς. Ε, ένα άλλο θέμα τώρα. Αρχίζει να αδειάζει η Μεσόγειος. Οι μη κυβερνικές οργανώσεις ε, σταμάτησαν να στέλνουν τα πλοία τους για αναζήτηση και διάσωση η επιχείρηση Σοφία παίρνει τέλος, ε, ε, υπάρχει ακόμα βεβαίως η, υπηρεσία, η, η, επιχείρηση Διτέμις ε, της Frontex όμως είναι 30 μίλια μακριά από τις ακτές μας, έτσι, 30 ναυτικά μίλια. υπάρχει όμως αυτή η επιστολή από την DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς εσάς που προτείνει μια συνεργασία μεταξύ Frontex και της υπηρεσίας ε, αναζήτησης και διάσωσης στη Λιβύη, των, των αρχών της Λιβύης. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε, σε μια άδεια Μεσόγειο, όπου υπάρχουν μόνο εμπορικά πλοία στην πραγματικότητα. Σας ζητείτε να πάτε εκεί κάτω τόσο νότια και θα συνεργαστείτε εκεί με τους Λίβιους ε, στα πλαίσια των δικών τους κανόνων και τα δικά τους κέντρα αντί για το κέντρο της Ρώμης ή δεν θα συμβεί τελικά κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή ποια θα είναι η δική σας, ο δικός σας ρόλος εκεί MRCC ε, λέγεται αυτό στη Λιβύη. Θα συνεργαστείτε μαζί τους ή με το κέντρο που υπάρχει στη Ρώμη. Ε, υπάρχει μια απόσταση, έτσι από το Θέμης, από την επιχείρηση θύμή στη Βόρεια Μεσόγειο και τη Λιβύη. Υπάρχει γεωγραφική απόσταση. Από πρακτική λοιπόν πλευρά αλλά και από νομική τελικά ποιο έχει την ευθύνη, ε, αν δηλαδή εσεί είστε το πιο κοντινό πλοίο στην περιοχή, ε, για να μια επιχείρηση διάσωση και σα ζητήσουν οι Λίβοι να κάνετε κάτι τέτοιο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριο Κολμέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Τραχά, ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα κύριε Λετζερή και να σας πω ότι όλοι οι υπάλληλοι που ήδη έχει προσλάβει η Frontex κάνουν όχι μόνο εξαιρετική δουλειά αλλά και δύσκολη δουλειά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Υποστηρίζω εξαιρετικά το γεγονός ότι αυξάνονται οι υπάλληλοι της Frontex με 10.000 προσωπικό. Προσικά είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός. Να κάνω όμως και μια ερώτηση η οποία δεν ε, έχει να κάνει απαραίτητα με τις ερωτήσεις που ήδη ακούσαμε. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς. Έχετε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε και θα έπρεπε να αλλάξει το νομικό πλαίσιο προκειμένου να σας επιτρέψει να διαμορφώσετε με πραγματικά αποτελεσματικό τρόπο την εργασία σας. Μπορούμε στην ε, θεωρία να αποφασίσουμε ότι θέλει άλλους 50.000 υπαλλήλους η Frontex. Σε κάποιο σημείο λοιπόν θα είχατε πάρα πολλούς υπαλλήλους. Το ερώτημα όμως είναι, θα επέλει αυτό πραγματικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της μετανάστευσης. Δεν το πιστεύω. Γιατί προφανώς χρειαζόμαστε να υπάρχουν απαρκείς υπάλληλοι στη Frontex είναι εξαιρετικά απαραίτητο να ε, μην πνίγεται κόσμο στη Μεσόγειο. Θέλουμε όμως να αποφύγουμε να έχουμε πληθώρα ε, προσωπικού για να καλύψουμε ουσιαστικά νομικές ελλείψεις, ε, τις οποίες τις καταχωρίζουμε, τις καταγράφουμε, αλλά δεν τις επιλύουμε. Άρα το ερώτημα είναι τι πρέπει να αλλάξουμε στο νομικό πλαίσιο προκειμένου πραγματικά να μπορούμε να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και έλεγχο του ποιο πραγματικά έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διατηρούμε και την ενόμη τάξη τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Χάουατς έχει τον λόγο. Κύριε Λετζέρη, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι απλό. Ε, δεν φτάσαμε εκεί την τελευταία φορά που είχατε έρθει. Αυτά, αυτός ο αριθμός των 10.000 ανθρώπων, των 10.000 προσωπικό, από πού προέρχεται. Είναι αίτημα της Frontex προς την Κομισιόν. Σας είπαν πόσους χρειάζεστε, χρειαζόμαστε 10.000. Και αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, από πού προέρχεται αυτός ο αριθμός. Και δεύτερον, ποιοι είναι οι βασικοί η δημοσιονομική για το 2020 και πού δέχεστε τη μεγαλύτερη πιέση σε δημοσιονομικό επίπεδο για το επόμενο έτος. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε για λίγο. Έχετε... Όχι, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Ναι, βεβαίως. Πολύ σύντομα. Από όσο θυμάμαι, αυτός ο αριθμός των 10.000 προέκυψε στην ομιλία του κυρίου Γιούνκερ για την κατάσταση τη Ένωση και μετά συμπεριλήφθηκε στο, στην πρόταση για το πολιτιστικο πλαίσιο. Σημείωσα τι ανησυχίε τη κυρία Γκρέσλε για το πώ θα κοστίσουν όλα αυτά. Ναι. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Μιντάου και... Ναι, μου το επιτρέπετε πρόεδρε να τελειώσω. Ήθελα λοιπόν εν συντομία να επιβεβαιώσω ότι μετά την ολοκλήρωση των πραγματεύσεων οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προετοιμάζουν ένα μια αναθεωρημένη δήλωση ε, σε ό,τι αφορά την, ε, τον οικονομικό αντίκτυπο της ε, συμφωνίας ε, αναέτος και ελπίζω αυτό να βοηθήσει την κυρία Γκρέσλε τις επόμενες μέρες θα συμβεί αυτό. Τις επόμενες μέρες. Και βεβαίως το τελευταίο μου σχόλιο σε ό,τι αφορά τον ε, συντελεστή διόρθωσης που εφαρμόζεται με μεγάλη λύπη η Κομισιόν σημείωσε ότι η πρότασή της να επιτρέψει μια αύξηση του συντελεστή για να φτάσουμε στα 100% δεν λήφθη υπόψη στην τελική συμφωνία εμείς πιστεύουμε αυτό θα έχει διευκολύνει πολύ τις δυνατότητες της υπηρεσίας ε, για να μπορέσει να ε, προβεί στις ε, προσλήψεις που πρέπει να κάνει και να πετύχει τους στόχους της. Μάλιστα, ευχαριστώ, ολοκληρώσατε. Και τώρα η διευθύντρια της DG Home. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Νομίζω όμως τα είπε ο συνάδελφος, ο κ. Σορέλο, οπότε δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω αυτά που είπε. Συνεργαζόμαστε στενά ε, στα πλαίσια των τελευταίων αυτών υπολογισμών και θα τα έχετε σύντομα. Θα είχα και εγώ δύο ερωτήσεις να κάνω, αν μου δίνετε τη δυνατότητα. Κύριε Γενικά, Γενική Διευθυντά, ε, τα κράτη και η Ευρώπη μήπως έχουν μπερδευτεί ε, σε κείμενα τα οποία νομικά κλπ. τα οποία είχαν ε, εκπονηθεί πριν από την μαζική μετανάστευση και αυτή την παγκοσμιοποίηση των μεταναστευτικών ροών. Μήπως μπορείτε να μας πείτε και ποιες είναι οι συστάσεις που θα μπορούσατε να μας δώσετε έτσι ώστε να τροποποιηθούν αυτά τα κείμενα για να μην είναι αναχρονιστικά. Δεύτερον, δημιουργία 10.000 θέσεων. Μήπως ε, με αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν ίσως να μελετήσουν για να ε, ε, αφαιρεθούν κάποιες από τις θέσει αυτές, δηλαδή κάποιες μετακινήσεις ενδεχομένως και από τους εθνικούς προπολογισμού προς τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ε, δέκα λεπτά επιπλέον θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα με την κατανόηση των διερμηνέων. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο όσον αφορά την διάσωση, έρευνα και διάσωση για τους λόγους στους οποίους ε, ήδη ε, εξηγήσατε Έχουμε περισσότερα ε, σημεία κοντά στις ακτές της Βόρειας Αφρικής ε, και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και κυρίως με το Δίκαιο της Θάλασσας ε, σε περίπτωση κινδύνου ε, έχουμε εναέρια μέσα τα οποία σε περίπτωση κατά την οποία έχουν διαπιστώσει περίπτωση κινδύνου πρέπει έχουν υποχρέωση παρέμβασης μέσω των όλων των μέσων θαλασσίων και λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας και μέσα από το συντονισμό του ε, Κέντρου Θαλάσσιου Εναερίου Συντονισμού. Επίσης έχουμε και ανάπτυξη MRCC και από την άλλη πλευρά της Μεσογείου αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει διαρθρωμένη διμερής ε, συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και την Λιβική MRCC. Όμως έχουμε ένα καινούριο project ε, που έχει στόχο ακριβώς την ανάπτυξη MRCC στην Τρίπολη γιατί πραγματικά ε, μπορεί να ελέγχει με τον τρόπο αυτό μια μεγάλη περιοχή της ε, Μεσογείου. Ε, οποτεδήποτε λοιπόν το ζήτημα είναι τι κάνουμε σε περίπτωση που διαπιστώσουμε μια κατάσταση κινδύνου και δεν υπάρχει maritime asset εκεί κοντά. Επίσης, βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, της υπηρεσίας ακτοφυλακής νορεφυλακής. Ε, ναι, βεβαίως πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Βεβαίως έχει βελτιωθεί ε, πάρα πολύ έχει βοηθήσει η υπηρεσία τα κράτη-μέλη 10% των ε, παρατύπων μεταναστών που έφτασαν ε, σε ευρωπαϊκές χώρες ε, επεστράφησαν στις αρχικές χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Πάντως πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και της υπηρεσία έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα ICT σε πραγματικό χρόνο. Και η πρόταση που έκανε η Κομισιόν ε, όσον αφορά την νέα οδηγία για τις επιστροφές πιστεύουμε ότι είναι προς, τον, προς την σωστή κατεύθυνση. Εμείς είμαστε παρόντες στα εξωτερικά σύνορα και ε, από τη στιγμή ε, που ε, έχουμε εκεί ε, μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να υποβάλουν αίτηση ασύλου ούτε νομιμοποιούνται για άδεια παραμονής θα πρέπει να επιστραφούν. Να σας υπενθυμίσω επίσης 5.000 συνοριοφύλακες λείπουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί καταλήγει η μελέτη αξιολόγησης. και σύμφωνα με τα κράτη-μέλη 110.000 θα έπρεπε να είναι οι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν δηλώσει τα, ε, ήδη ε, τα κράτη-μέλη. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσες είναι οι ανάγκες, καταλαβαίνετε τι αντιπροσωπεύει το, το σύνολο αυτό των 10.000 ε, υπαλλήλων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Τώρα, για τον προπολογισμό 2020, να πω ότι τώρα βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο. Την προηγούμενη εβδομάδα εγώ ε, υπέβαλα στο Δυτικό Συμβούλιο τους, ε, τα περσινά στοιχεία Ξέρω, ξέρω ότι είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να προσαρμοστούμε και να ξανα... ίσως θα πρέπει να ξαναπευθυνθώ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν ε, ε, διαπιστώνω να υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος ε, για το 20 αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να προσαρμοστούμε μετά από τη μεταβατική περίοδο. Αλλά αυτό αυτό, αυτά τα λέμε βασιζόμενοι ε, στο, στα τρία χρόνια πριν. Όσον αφορά τις δικές σας ερωτήσεις κύριε Πρόεδρε, κατά πόσον είναι αναχρονιστικά ε, τα κείμενα τα οποία έχουμε τώρα στη διάθεσή μας πέρα από την μετανάστευση υπάρχει το, το θέμα της κινητικότητας. Είναι παγκοσμιοποιημένη η κατάσταση ε, και βρισκόμαστε, ζούμε σε μια χώρα όπου άνδρες, σε μια κατάσταση όπου άνδρες, γυναίκες, εμπορεύματα κινούνται, κυκλοφορούν. Επομένως θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή και να αντιμετωπίσουμε βέβαια και το πρόβλημα και της απομάκρυνσης των παρατύπων μεταναστών από την άλλη μεριά. Θα πρέπει ε, να δώσουμε όλες τις ε, δυνατότητες ε, ναι, των, της νόμιμης διάσχεσης συνόρων. 700 εκατομμύρια νόμιμες διελεύσεις ε, ε, συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κάθε χρόνο και επομένως θα πρέπει να ελέγχονται όλες αυτές οι διασχίσεις Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνεται όλο και πιο εύκολη διάσχεση των συνόρων για ανθρώπους που έχουν το δικαίωμα να τα διασχίσουν. Επομένως εταιρικέ σχέσεις έτσι ώστε να αποτελέσει, να συνεχίσει να αποτελεί η Ευρώπη ε, έναν χώρο ανταλλαγής ε, πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Και για τη Λιβύη τι έχετε να μας πείτε? Ε, la Για τη Λιβύη, ναι, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά την συνεργασία. Έχουν ληφθεί αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργηθεί ε, και λιβική ε, ε, συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. 46 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για αυτήν την δραστηριότητα, όμως επιχειρησιακές άμεσες ε, επαφές όσον αφορά την οργάνωση δεν έχουμε εμείς. Εμείς ενεργούμε ε, αυτό μάλλον γίνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και εμείς συμμετέχουμε στην κατάρτιση των ακτοφυλάκων της Λιβύης. Πρόσφατα έγινε μια τέτοια, ε, ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάρτισης ε, επίσης ε, και στην η αστική Γιούμπαμ Λίμπια που είναι η αστική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Λιβύη έχει αναλάβει ε, τέτοιου είδους ε, καταρτήσεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά αλλά και το προσωπικό σας που κάνει τόσο ευαίσθητη δουλειά και την αναγνωρίζουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ επίσης τους εκπροσώπους των Επιτροπών Κοντ και Λίμπε. Ευχαριστώ και τους αντίστοιχους προέδρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ευχαριστούμε την Κομισιόν και κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που μας έδωσαν αυτόν τον παραπάνω χρόνο και είχαμε διερμηνία πέρα από τις κανονικές, τις κανονικές τους ώρες εργασίας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ. Στην ίδια έφερα.